στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η έκθεση Κράμερ, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Τεχνολογία των Μεταφορών για τη βιώσιμη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη. Τον λόγο έχει ο εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, είχαμε καλά αποτελέσματα και ε, μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή. Η έκθεση πρωτοβουλία είναι αντίδραση στην ανακοίνωση της Κομισιόν για την έρευνα και την καινοτομία για την μελλοντική ε, κινητικότητα στην Ευρώπη για την ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής. Συμφωνήσαμε όλοι πως οι καινοτομίε ε, μέχρι στιγμή δεν απαρκούν και πρέπει να βελτιωθούν. Στόχος της έκθεσης είναι να συμβιβαστεί η ερευνητική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους μας. Δεν θέλουμε παραδείγματο χάρη να επαναλαμβάνεται η έρευνα. Πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν ευκολότερα να λάβουν ευρωπαϊκά κονδύλια και βέβαια να ενισχύσουμε τα διασυνοριακά έργα. αλλιώς θα καταλήξουμε με ένα μοσαϊκό και τα κενά υπάρχουν ακριβώς στα σύνορα, δηλαδή ε, η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία δεν υπάρχει ακόμα μετά από 20 χρόνια και βεβαίως χρειάζεται να δούμε το τι εννοούμε καινοτομία. Δεν είναι μόνο τεχνολογική καινοτομία, αλλά και η συμπεριφορά των ανθρώπων πρέπει να αλλάξει. Γιατί πλέον βλέπουμε πως η κατοχή του αυτοκινήτου δεν είναι το σημαντικό όπως το δεκαετία του 50 και 60, αλλά σημασία έχει η χρήση του. Πώς μπορούμε να τα επιτύχουμε αυτά. Πολιτική ουδέτερη ως ε, προς την ε, τεχνολογία πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε ένα κομμάτι. Π.χ. το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει μόνο πλεονέκτημα εάν δούμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Παραγωγή, χρήση και ανακύκλωση. Και εκεί πέρα... Ε, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πίσω από τα συμβατικά αυτοκίνητα. Γι' αυτό λέμε πως είναι σημαντική η ουδετερότητα της τεχνολογίας μας. Ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, όχι το πώς θα φτάσουμε εκεί. Γιατί εγώ μηχανικός δεν είμαι. Και το ίδιο δεν ήταν ε, βεβαίως ε, και οι σκιώδησίδες. Επιπλέον πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει το παράδειγμα η δική μας υπηρεσία πρέπει να κινηθεί με τρόπο πιο βιώσιμο, δηλαδή με αυτοκίνητα τα οποία θα καταναλώνουν λιγότερο και θα κάνουν λιγότερο θόρυβο. Θέλουμε επίσης να έχουμε μια βάση δεδομένων για, στο, για λόγους διαφάνειας και σημαντική επίσης είναι να υπάρξει μια ολοκλήρωση, να πηγαίνει κανείς με τα πόδια, με το ποδήλατο, με τις συγκοινωνίες, με το αυτοκίνητο και αυτά να συνδυάζονται. Και όχι απλά να κοιτάμε πώς θα πάμε από το α στο β, αλλά να δούμε από πόρτα σε πόρτα πώς θα φτάσουμε. Εκεί πέρα πρέπει να αξιστεί η αποτελεσματικότητα. Υπάρχει λοιπόν ευρεία συνένεση, είχαμε μεταξύ μας, πως ε, πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτά. Και ιδιαίτερα χαίρομαι για το ότι υπήρξε με τη συμφωνία στη μείωση του θορύβου, κάτι το οποίο δεν ίσχυε πριν από 2-3 χρόνια, γιατί ξέρουμε πως ο σιδηρόδρομος θα έχει μέλλον στην Ευρώπη μόνο αν αντιμετωπίσει το πρόβλημα του θορύβου. Και με κάποιες μελέτες είδαμε πως ε, 2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για, τα, για το τροχαίο υλικό μπορούμε να μειώσουμε τον θόρυβο των σιδηροδρόμων στο μισό, ειδικά στον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές. Και έτσι έχουμε μια κατάσταση που οποία είναι μηδέα υποφελής. Αυτά και σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Έχω τέσσερις ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μπάνκι. Elnök úr, a jelentésből két pontot szeretnék kiemelni, ahhoz szeretnék hozzászólni. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα δημόσια μέσα μεταφοράς, θα πρέπει σαφώς να αναπτύξουμε κόμβους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές έτσι ώστε να μειωθεί η μόλυνση της ατμόσφαιρας, τα πλήγματα στο περιβάλλον ενισχύοντας μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα είτε ηλεκτρικά λεωφορεία κτλ. Δεύτερον, θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε την πλευρά της ασφάλειας αυτών των μεταφορικών μέσων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Κάτι που θα πρέπει να επιστρέψει και στο κέντρο των πόλεων μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νταντσίλα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι βιώσιμες μεταφορές απαιτούν να κατανοούμε και τα διάφορα στάδια στην αλυσίδα μεταφοράς ε, στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Για να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε τις διαφορές μας και για να βελτιώσουμε την κινητικότητα θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε διαπεριφερειακές συνδέσεις και ε, συνδέσεις ε, στα σύνορα. Ένα σύστημα παρακολούθησης για την έρευνα και την ανάπτυξη στι μεταφορές ε, θα είναι προ όφελο όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται τακτικά ε, δωρεάν πληροφορίες ώστε να μπορούν να δώσουν και κατάλληλα τι επιδοτήσει. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κράμερ, σας ευχαριστώ για το έργο σας, ευχαριστώ για το όσα έκανε η ομάδα σας και για την ε, συνεργασία σας. Ήταν ε, χαρά να συνεργαστούμε σε αυτή την έκθεση για τις ευφύης μεταφορές, διότι θεωρώ ότι αποτελεί κλειδί για τις αλλαγές ε, στην οτροπία των Ευρωπαίων πολιτών προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε και τη συμμετοχή των χρηστών και τη ε, συμμετοχή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε ένα μηχανισμό ο οποίος θα έχει ένα καλύτερο μελλοντικό σχέδιο μεταφορών ώστε να αλλάξουν οι κατάλληλες νοοτροπίες και να δώσουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία. Οι τοπικέ και περιφερειακές αρχές ε, αντιμετωπίζουν με μεγάλο ποσοστό κοινοτομία τα προβλήματα τη καθημερινή κοινότικότητα που αποτελούν πρόβλημα για του πολίτε καθημερινά. Και η συνεργασία του ήταν χρήσιμα για να μπορέσουν να αλλάξει το πλαίσιο και να αλλάξει η νοοτροπία. Ζητάμε επίση και τη συνεργασία από τι κατάλληλε αρχέ, διότι η καινοτομία προχωρά πολύ πιο γρήγορα από τι διοικητικές διαδικασίε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουν μια πιο ανοιχτή στάση για να μπορέσουν να δώσουν κατάλληλε και για τα οι οχήματα, αλλά και για τα ποδήλατα, τα δίκυκλα και γενικώ ηλεκτρικά οχήματα. Ευχαριστώ, ο κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καινοτομία είναι καθοριστική, όπως διαβάζουμε και στην έκθεση, για να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στα μέσα μαζικής ε, μεταφοράς. Στην έκθεση βλέπουμε την περιγραφή της κατάστασης σε πολλές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, την αποδυνάμωση των ε, δημόσιων μέσων μεταφοράς, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται στη χώρα μας από μέρους της Τρόικας. Η αποτελεσματικότητα μειώνεται κατά 20%, η ταχύτητα αύξηση των τιμών είναι πασιφανής και ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι χρήστες επιστρέφουν στα ιδιωτικά οχήματα και αυτό είναι τραγικό. Βλέπουμε επίσης ότι οι συστάσεις οδηγούν προς ε, μια βιώσιμη στήριξη των μέσων μαζικής ε, μεταφοράς, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίφαση με τα πραγματικά μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ρέντινγκ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Κράμερ, τον εισηγητή, καθώς και την Επιτροπή Μεταφορών, αλλά και την Ολομέλεια για την στήριξη στην πρόταση της Επιτροπής πρόκειται για μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για μας η καινοτομία στα μαζικά μέσα μεταφορών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις μεταφορές αλλά και για την υλοποίηση των στόχων μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όσον αφορά τις συστάσεις και τις προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τις εξετάσει προσεκτικά και σίγουρα θα υιοθετήσει πολλές από αυτές γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι οι προκλήσεις στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας έτσι ώστε να αναπτύξουμε συστήματα για περισσότερη κινητικότητα, πιο ασφαλή μεταφορά και εδώ βεβαίως χρειάζεται μια προληπτική δράση. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι προτάσεις σας θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Η συζήτηση τελείωσε. Η ψηφοφορία αύριο στις 12 η ώρα. Επόμενο θέμα. Έκθεση της κυρίας Κλέβα και εφαρμογή και αντίκτυπο των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και